Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε με τις επεξηγήσεις ψήφου. Είναι το επόμενο σημείο στην ημερήσια μας διάταξη. Θα ξεκινήσουμε με τη σύσταση Κριστιαν Πρέντα. Η κυρία Μακόβε έχει το λόγο. Μακοβέη. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί